President. Ach Gott. okay, David. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα να σας παρακαλέσω να καθίσετε. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ε, έχουμε την ψηφοφορία με απλουστευμένη διαδικασία για την έκθεση της κυρίας Φιγκερέντο. Το λόγο έχει η συγγήτρια. Παρακαλώ, συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα